Η χθεσινή εκδήλωση αφορούσε σε ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας και είχε μια ιδιαίτερη σημασία γιατί οφείλεται στην ενεργοποίηση κυρίως των Ευρωπαίων βουλευτών, ε, πολιτών. Έγινε για να υποστηρίξει όσο μπορεί το πανευρωπαϊκό κίνημα Right to Waters, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση σχετικού ψηφίσματο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το γεγονό ότι στη σημερινή συγκυρία, που κινδυνεύουν όσα ανθρώπινα δικαιώματα έμειναν αλόβητα, ο ενεργός ρόλος του πολίτη σήμερα προβάλλει κυρίαρχος και απαραίτητος αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την τραγική πραγματικότητα την οποία οι κυρίαρχες δυνάμεις διαμορφώνουν εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα και το ότι επίσης το κίνημα απέδειξε ότι η κοινή δράση έχει αποτελέσματα για τις αξίες που αφορούν στην ποιότητα και την ε, καθημερινότητά μας και την αξιοπρέπειά μας. Στη σημερινή πραγματικότητα που 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και πάνω από 2,6 δισεκατομμύρια, περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό είναι βασικό χαρακτηριστικό του κύκλου της φτώχειας που ε, κτυπά αυτές τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο και η αδυναμία της αντιμετώπισης του οδηγεί σε παγκόσμια ανισότητα και αδικία. Οι αυξανόμενες τάσεις για εμπορευματοποίηση του νερού, η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η άνηση παροχή υπηρεσιών, η έλλειψη δίκαιων, βιώσιμων και υπεύθυνων πρακτικών είναι όλα άμεσες αιτίε της σημερινής παγκόσμιας κρίσης. Το νερό λοιπόν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και αναπαλωτρίο το κοινωνικό αγαθό και όχι απλά μια πρώτη για εμπορική χρήση και επειδή στο μέλλον θα γίνει το πιο πολύτιμο αγαθό και η πίεση θα αυξηθεί. Εμείς, σαν πολίτες, δεν πρέπει να, να, οπισθοχωρήσουμε. Πρέπει να εντείνουμε τις δράσεις μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι σε αυτόν τον πλανήτη δικαιούνται και θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το φυσικό αγαθό. Ε, πριν δώσω τον ε, λόγο στους ε, κυρίους παρισταμένους, που είναι οι κύριοι βουλευτές οι οποίοι στηρίξαν την ε, αυτή την εκδήλωση και οι καλεσμένοι μας. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και συνέδραμα στον επιτύχει αυτή η εκδήλωση. Ε, θα σας αναφέρω ε, ε, επιγραμματικά τα, τα, τα συμπεράσματα, που το πρώτο είναι ότι η αντίληψη που επικρατεί αυτή τη ε, στιγμή στους Ευρωπαίου πολίτες είναι ότι το νερό είναι δημόσιο, συλλογικό και κοινωνικό αγαθό και απαιτείται η εξασφάλιση της πρόσβασης του σε όλους τους πολίτες το δεύτερο είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε νομοθετική διαδικασία, να υλοποιήσει ε, τις ρητές προβλέψεις του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε με την, με την γνωστή πρωτοβουλία Right to Waters από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τρίτον ότι έχει γίνει συνείδηση σε όλους ότι πρέπει να υπάρξει μια διευρυμένη πανευρωπαϊκή συνεργασία που θα μπορεί να στηρίξει τόσο αγώνες και διεκδικήσει σε εθνικό επίπεδο, αλλά και να πιέσει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν προς αυτό. Θα δώσω το λόγο αμέσως στους συναδέλφους για πολύ μικρές τοποθετήσεις του ενός λεπτού θα παρακαλούσα, στον κύριο Λόπες καταρχήν Uh, Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο, διότι συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα υπόθηκαν χθε ε, κατά τη διάρκεια τη εξαιρετική πρωτοβουλίας που είχαμε εκ μέρους του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού κόμματο ε, θεωρούμε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και του σχετικού μοντέλου μέσα στο οποίο ζούμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε έξαρση των ιδιωτικοποιήσεων. Μανία με τις ιδιωτικοποιήσεις θα το έλεγα έτσι. Ε, που χαρακτηρίζει πλέον πολλούς τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και φυσικά το νερό είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Αυτό οδήγησε, όπως υπόθηκε χθε, σε αύξηση του κόστους για τους ανθρώπους, στην υποβάθμιση των υπηρεσιών, στον περιορισμό της πρόσβασης στο νερό για πολλές μερίδες του πληθυσμού, ειδικότερα για τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τις αστικές περιοχές. με σημαντική επίπτωση στο κόστος για τον ε, γενικότερο πληθυσμό φυσικά. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, ένα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπου εργαζόμαστε, γνωρίζουμε ότι καμία νομοθεσία συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναφέρει ότι υπάρχει υποχρέωση ιδιωτικοποίησης του νερού. Κανείς δεν λέει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν ε, διευθετηθεί έτσι ώστε η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός των κυβερνήσεων να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και πολλές είναι οι αντικρώμενες φυσικά πολιτικές ε, ε, εντός της ενιαίας αγοράς. Ε, το ελεύθερο εμπόριο κτλ. Και όλα φυσικά αυτά αντιμάχονται τις ανάγκες των ανθρώπων. Ένα από τα πράγματα που υπόθηκαν χθες ε, για να συνοψίσω και να κλείσω σύμφωνα απόλυτα με την ε, ανάγκη να υπάρχει ένα οικουμενικό δικαίωμα για το νερό και συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη διαχείρισης των υδατινών πόρων ξεχωριστά από τους νόμους της αγοράς. Ε, ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας και να μεριμνήσουμε ώστε να παραμείνει δημόσια η διαχείριση του νερού. Αυτά για μας ε, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση ε, και να βελτιωθεί ο μαζικός αγώνας ώστε να επανακτήσουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε ε, την ιδιωτικοποίηση του νερού, την οργάνωση φυσικά των εργαζομένων και του πληθυσμού, διότι χωρίς ε, μια τέτοια οργάνωση δεν θα καταστεί ε, δυνατή ο σωμαζικός αγώνας αλλά και η απόλυτη ανάγκη για πολιτικές αριστερού χαρακτήρα οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν φυσικά από αριστερές κυβερνήσεις αλλά όχι μόνο αριστερές ε, στα χαρτιά, ε, να είναι αριστερές ε, κυβερνήσεις που πράγματι υλοποιούν πολιτικές οι οποίες ευθυγραμμίζονται και συμμορφώνονται με τις ανάγκες των λαών και για το συμφέρον των χωρών. Εδώ θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ. Πολύ πολύ σύντομο. Um, θα είμαι σύντομη Σύμφωνο με όσα είπατε για τι ιδιωτικοποιήσει και το μήνυμα που θέλω να στείλω σήμερα είναι προ την Κομισιόν και κυρίω προ τον Επίτροπο Βάλε ως εισηγήτρια τη έκθεση που πέρασε το Σεπτέμβριο του 2015 που εκφράζει το σαφέ αίτημα της Κομισιόν να αναγνωριστεί ένα οικομενικό ε, δικαίωμα στο νερό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Κομισιόν όμω δεν αποκρίθηκε σε αυτή την έκθεση, όπω δεν αποκρίθηκε στην πρωτοβουλία των πολιτών και η αλαζονία τους ως προς τη δημοκρατική διαδικασία μας δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες, ειδικότερα για ένα κοινωνικό ζήτημα όπως το νερό, καθώς και η υποκρισία των δράσεών τους, όταν λένε ότι κρατούν ουδέτερη στάση όσον αφορά το πώς οργανώνουν τα κράτη-μέλη το, ε, ε, τους υδάτινους πόρους, τα εστιαστήκαμε στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι η Τρόικα ε, προωθεί την ατζέντα της ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα και στη χώρα μου στην Ιρλανδία έχουν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία διότι δεν έχουμε ε, Φορά αλλά μια γενική φορολογία οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί το προϊόν για να γίνει ιδιωτικοποίηση οπότε αναγκάζουν την εγκατάσταση μετρητών νερού παρότι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μετρητές δεν είναι αποτελεσματικοί και δεν οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης νερού όπως ισχυρίζονται. Αυτό το μήνυμα ήθελα να στείλω σήμερα για την Κομισιόν και για τον Επιτροποβέλα ε, πρέπει να ακούσει τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσει να παραβλέπει τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος, όπως ε, είπα και χθες. Το νερό είναι ένα από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους ε, του πλανήτη μας. Χρειαζόμαστε το νερό όπως χρειαζόμαστε τον αέρα για να αναπνέουμε. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε καθαρό και προσιτό ε, πόσιμο νερό και σε αποχέτευση. Και επειδή ο παγκόσμιος πληθυσμό αυξάνεται πάρα πολύ, επειδή υπάρχει μόλυνση των ε, επιφανειακών εδάτων από τη γεωργία και τη βιομηχανία, το νερό είναι πολύ περιορισμένος πόρος. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι στα χέρια διεθνών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε τώρα. Αυτή είναι η επιθυμία των πολιτών. Και υπάρχει επίγουσα ανάγκη δράσης από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις για την πολιτική. Μόνο οι πολιτικοί, αυτοί που καθορίζουν την πολιτική, μπορούν να διασφαλίσουν το δικαίωμα σε καθαρό και σε προσιτή τιμή νερό για τον πληθυσμό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εθνικές ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομικές, ε, συγγνώμη, νομοθετικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το νερό και η διαχείρισή του να παραμείνει ή να επανέλθει στο δημόσιο τομέα. Είναι απόλυτα αναγκαίο να καταπολεμήσουμε την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού. Θέλουμε κοινή δράση για να συνεχιστεί ο αγώνας για το ανθρώπινο δικαιώμα πρόσβαση στο νερό και εντός και εκτός, του Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την πίεση όλοι από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με δίλεπτε τοποθετήσει, μου επιτρέψετε να πω, από την μοναδική κυρία που είναι πάνω στο πάνελ, την κυρία Κανελοπούλου πρώτα, που είναι από το Save Creek Water, και μετά θα πάμε στου κυρίε. Ε, δεν ξέρω αν πρέπει να, διαβάσουμε τώρα το ψήφισμα που εξεδόθη. Ναι. Ε, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διήμερη διαδικασία ε, συγκεντρωθήκαμε εδώ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού, εκπρόσωποι συνδικάτων, επιστημονικών φορέων και κινημάτων από πολλές χώρες της Ευρώπης. Επισημαίνουμε από κοινού ότι την ίδια στιγμή που στα κέντρα λήψης αποφάσεων στη Γαλλία και στη Γερμανία το νερό επαναδημοτικοποιείται ύστερα από την αποτυχία του μοντέλου ιδιωτικοποίησης που προωθήθηκε επί δεκαετίες από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Δέλτα ζητείται από τις χώρες υπό οικονομική επιτήρηση, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ίδρυυσης και μάλιστα κατά παράβαση τόσο της ουδετερότητας της Κομισιόν, όσο και του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Right to Water. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείε ίδρυυση και αποχέτευση Αθήνα και Θεσσαλονίκη ορίστηκε ω μνημονιακή υποχρέωση να ενταχθούν στο νέο Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων. Παράλληλα, άδειασαν τα ταμεία των διαθεσίμων της ΕΙΔΑΠ με επανειλημμένες κινήσεις επιστροφής κεφαλαίων και επενδύσεων ύψους 77 εκατομμύριων ευρώ, την ώρα που ζητείται από το Asset Development Plan να πολυθούν το 11% της ΕΙΔΑΠ και το 23% της ΕΙΑΘ. Ζητούμε τη συμμόρφωση όλων των εθνικών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών οργάνων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και τις δικές τους διατυπώσεις, ότι το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2060. Ζητούμε να συμμορφωθούν επίσης με τις δημοκρατικά εκφρασμένες μέσω δημοψηφισμάτων απόψεις των ευρωπαϊκών λαών, όπως στην Ιταλία, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, που έχουν καταδικάσει επανειλημμένα την έμεση ή άμεση ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού και της διαχείρισής του. Θέλουμε να τονίσουμε ακόμη ότι οι υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να είναι κερδοφόρες, να είναι στην πέμπτη θέση εφαρμογής της οδηγίας σε θέματα αποχέτευσης, με συνέπεια η Ελλάδα να είναι τρίτη στην Ευρώπη σε καθαρότερες ακτές. Παρέχουν επίσης εξαιρετικό ποιοτικό νερό σε ένα από τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ευρώπη προσφέροντας κατά περιπτώσεις κοινωνικά τιμολόγια για τους οικονομικά ασθενέστερους. Σε συντονισμό με τους φίλους μας του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού από όλες τις χώρες, το επόμενο διάστημα όλοι οι συνυπογράφοντες θα ασκήσουμε πίεση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται δράσεις νομικές, συνδικαλιστικές, καμπάνιες τοπικής και εθνικής εμβέλειας και γενικότερα δράσεις στο πλαίσιο του κάθε φορέα. Παραδειγματικά μόνο αναφέρουμε, πρώτον, μέλη του ΣΕΙΠ έχουν ζητήσει με επίσημο έγγραφο τη δημοσιοποίηση κάθε επικοινωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των ελληνικών κυβερνήσεων μετά την 24η Μαΐου 2014 και τη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορούν την ένταξη των ελληνικών υπηρεσιών ίδρυυσης στο υπερταμείο. Δεύτερον, στις 20 Μαρτίου εκδικάζεται η προσφυγή των μελών του ΣΕΚΕΣ σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της ΕΙΔΑΠ για επιστροφή κεφαλαίου ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που καθιστά αβέβαιο το οικονομικό μέλλον της εταιρεία. Τρίτον, προσφυγή έχουν καταθέσει και εργαζόμενοι της ΕΙΑΦ, καθώς πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με κάθε ένδικο μέσο κατά τη ένταξη των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ του υπερταμείο. Και φυσικά η Ομοσπονδία Εργαζομένων στι δημοτικέ επιχειρήσει Ήδρευση και αποχέτευση στην Ελλάδα χρηματοδοτεί ντοκιμαντέρ για την κατάσταση και το έργο των επιχειρήσεων αυτό, καθώ και τι αρνητικέ επιπτώσει τη ιδιωτικοποίηση σε δημοτικό επίπεδο παγκοσμίω. Επίση, τοπικά κινήματα όπω τη Χαλκιδική, τη Θάσο, την Κόρινθο, την Κρήτη έχουν ξεκινήσει συντονισμένες καμπάνιες ενημέρωσης πολιτών και δράσεων. Συμπερασματικά, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε πολιτική που μετατρέπει το νερό από κοινό αγαθό σε εμπόρευμα, συμπεριλαμβανομένης και της τάσεως ανάκτησης πλήρους κόστους, που σύμφωνα με επιστημονικούς φορείς δεν είναι εφαρμόσιμη. Ζητούμε από το Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσει να στηρίζει τους αγώνες μας και να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών στο θέμα αυτό, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεσμών, που βρίσκονται και δικαίως υπό έντονη αμφισβήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο. Πονδίας ναι. ΕΙΔΑ, τον, ναι, τον εργαζομένο στην ΕΙΔΑΠ. Ε, θα παρακαλούσα μονάχα στο δίλεπτο για να προλάβουμε να έχουμε και μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ε, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιώργο Συνιέρη, ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Εργαζομένων τη ΕΙΔΑΠ. Στο πάνελ εκπροσωπώ επίση και την εταιρεία τη ίδρυυση τη Θεσσαλονίκη, την ΕΙΑΘ, αλλά και όλη την, την Ομοσπονδία όλων των δημοτικών φορέων του νερού τη Ελλάδο. Ε, οπότε μιλάω εκ μέρου και των τριών που εμεί έχουμε ε, άτυπα δημιουργήσει τον κλάδο του νερού τη Ελλάδο. Συνδικαλιστικά εννοώ. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι στην Ελλάδα οι υπηρεσίε ίδρυυση και αποχέτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε παρέχονται από δημόσιους ή δημοτικούς φορείς. Στο λεκανοπέδο τη Ατική, η δημοτικου φορει στο λεκανοπεδιο τη αττικης η εταιρεια ιδρυυση και αποχέτευση πρωτεύουσα είναι η ΕΙΔΑΠ, έχει την αποκλειστική αρμοδίδα τη υδροδότης αποχέτευση και επεξεργασία λιμάτων και έχει στην ιδιοκτησία τη τα δίκτυα και τι εγκαταστάσει. Στη Θεσσαλονίκη, αρμόδια είναι η Εταιρεία Ίδρυυση και Αποχέτευση Θεσσαλονίκη, η λεγόμενη ΕΙΔΑΠ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι κατά δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση και αποχέτευση ΔΕΙΑ. Όπω καταλαβαίνουμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το νερό και ο κύκλος του νερού διαχειρίζεται καθαρά από το δημόσιο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του δημοσίου. Η θέση μας είναι αυτή, είναι απαράβατη. Ο αγώνας μας είναι και όλες οι προσπάθειες που κάνουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε κυβέρνηση οποιασδήποτε χώρα πρέπει στατηγική ε, σημασία συγγνώμη, πηγές πλούτου ε, γη τη να τι έχει στα χέρια τη και να τι ελέγχει η ίδια. Δεν είναι δυνατόν και είναι αδιανόητο εν ώψη μια κρίση που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα να προσπαθούν κάποιοι να εκμεταλλευτούν και να πάρουν όλη την περιουσία τη συγκεκριμένη περίπτωση του ελληνικού λαού και μάλιστα για 99 χρόνια. Εμεί είμαστε εντελώ αντίθετοι, θεωρούμε ότι τα κοινωνικά αγαθά και ειδικά όπω είναι το νερό πρέπει να παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου και οι αγώνε μα θα είναι μαζί με όλη τη συμμαχία γι' αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα σε ερωτήσεις. Δεν άκουσα. Τελειώσαμε, θα μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Έχουμε έρθει άλλους δύο. Λοιπόν, ε, μιλήσατε ως βουλευτής. Μέσα σε ένα λεπτό τα είπατε όλα, κύριε Σινιώρη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπέρι, εκπρόσωπο του ΣΕΚΕΤ για δημόσια ΙΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας, επίσης για ένα λεπτό για ένα Αυστηρά για ένα λεπτό. Ε, η μάχη για την κατοχήρωση της καθολικής, ατομικής και συλλογικής προσβασιμότητας σε επαρκές καθαρό πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης είναι θεμελιώδης προϋπόθεση του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο, είναι ο έμπρακτος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και είναι ο δρόμος να δημιουργήσουμε μια ισχυρή συμμαχία εργαζομένων και κοινωνίας για την υπεράσπιση του δημόσιου νερού. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε στο συμμετοχικό ενωτικό κίνημα εργαζομένων και συνταξιούχων και θα δώσουμε τη μάχη μαζί με όλα τα κινήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και το λόγο έχει ο κύριος Κακλής, Τριαντάφυλλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων. Για ένα λεπτό. ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό το θέμα και πολύ σύντομο. Σαν Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων εκφράζουμε την αντίθεσή μα σε οποιαδήποτε εμπορευματικοποίηση του νερού, ξεκινώντα από, από την ίδια την Οδηγία 2060 για τα νερά, όπου η πρώτη θεώρηση ε, αναφέρει ότι το είδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπω όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τη χάνει από κατάλληλη μεταχείριση. Ε, είναι ζωτική σημασία σαν αγαθό για τον άνθρωπο και συνοπτικά, σαν σύλλογο, οι πάγιε μα θέσει είναι ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό, απαραίτητο για την ύπαρξη ζωή και η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλέ, καθαρό και φθηνό νερό, καθώ και σε ποιοτικέ υπηρεσίε αποχέτευση είναι ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο οικονομική αποτίμηση και εμπορική δραστηριότητα. Οι υπηρεσίε σύνδρευση και οι υποδομέ εξασφάλιση νερού διαφόρων χρήσεων μπορούν να κοστολογούνται και να τιμολογούνται, αλλά δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε οποιοδήποτε τύπο ιδιοκτησία επί πόρων τη χώρα μα. Καλούμε την κυβέρνηση να μην απελευθερώσει την αγορά υπηρεσιών ίδρυυση και αποχέτευση, να, μην συμπεριλάβει τι υπηρεσίε ίδρυυση και αποχέτευση σε κανένα είδου εμπορικέ ή δανειακέ συμφωνίε. Τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση δημοσίων εταιριών ίδρυυση και αποχέτευση, όπω η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, πρέπει να αποσυρθούν από κάθε είδου συζήτηση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρέσει τον τομέα των υδάτων από την οδηγία για την απελευθέρωση, όπω άλλωστε έχει επανειλημμένα δεσμευτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση προς τους κυρίους. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ερμηνεύεται το αντιφατικό γεγονός που αναφέρατε ότι ενώ στους Δήμους των ε, ισχυρών κέντρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Παρίσι, Κάρδη ή το Βερολίνο προχωρούν σε επαναδημοτικοποιήσεις των υπηρεσιών γύρω από το νερό, οι Δήμοι των μικρότερων χωρών οθούνται προς την ιδιωτικοποίησή του. Ποια είναι η ερμηνεία που έχετε σε αυτό το γεγονός και επίσης πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η υποκρισία που αναφέρθηκε προηγουμένως στη στάση της Κομισιόν. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και να γίνει μια απάντηση γιατί περνάει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε. Παρακαλώ. Όχι, όχι, η κυρία που είναι πίσω σας. Sorry. Uh, Odil Harvey from... Uh, um, uh, από το Magazine που ε, στο Παρίσι. Μια διευκρίνηση. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία από την Ιρλανδία για ποιο λόγο, αν κατάλαβα καλά, είστε κατά των μετρητών νερού. Αυτό είναι μία μου ερώτηση. Ε, και τώρα στις διάφορες χώρες ε, εκφράζονται ανησυχίες ε, για το πόσο η αποχέτευση σχετίζεται με το νερό ή είναι ξεχωριστή. Ποιες είναι οι απόψεις σας γι' αυτό. Ίσως στη συνεδρία σας να το αναφέρετε, δεν ξέρω, έχετε κάποιους πίνακες που να απεικονίζουν την κατάσταση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες διότι δεν έχουμε μόνο την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία που εκπροσωπούνται εδώ. Θα ήταν καλό να δούμε την κατάσταση και στις υπόλοιπες χώρες. Να έχουμε περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιο που θέλει να κάνει. Παρακαλώ. Σκαρίμπα ε, Θήμιος λέγομαι, εκπροσωπώ την Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου ε, τον απλό πολίτη δηλαδή, χωρίς εξειδικευμένε γνώσεις και ο οποίος τώρα ενημερώνεται. Ε, μιλάμε για κίνδυνο ιδιωτικοποίηση του νερού. Είναι σήμερα σε εξέλιξη το νερό στην Ελλάδα, τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά τα τελευταία χρόνια μα βάλαν και δηλώσαμε μέχρι και το πηγάδι του, στο, του, του, στο χωριό του παππού. Το πηγάδι το δικό μα που το θεωρούσαμε παραδοσιακό δικό μα. Και το δηλώσαμε και αυτό σαν πηγή νερού. Ε, μπορείτε να μου πείτε με απλά λόγια, ποιο νερό που χρησιμοποιώ εγώ σήμερα με μια προσιτή τιμή ή, με, ή δωρεάν από το ποτάμι ίσως ε, θα πρέπει να το πληρώνω μετά την ιδιωτικοποίηση ακριβά γιατί η ιδιωτική εταιρεία έχει κατά κανόνα και αποδεκτά μόνο σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Το νερό της βρύσης, του πεγαδιού μου, του δικού μου, του προπάπου μου, ε, το νερό του ποταμιού για να αρδεύσει ο αγρότης το χωράφι του. Ευχαριστώ πολύ πολύ σύντομα γιατί ε, πρέπει να παρακαλέσουμε τους ε, κυρίους μεταφραστές αν μπορούν να μας δωσουν δυο δύο-τρία λεπτά ακόμη. Μια πρόταση είναι. Ε, Μα το ράξαμε από το ΣΕΚΕΣ. Υπήρξε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία τη Ελλάδο για τη μη ιδιωτικοποίηση για τη μη της ΕΙΔΑΠ και την επιστροφή των μεταχών στο δημόσιο. Έχει υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και αν όχι γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω το λόγο καταρχήν στην κυρία Κανελοπούλου για να απαντήσει την πρώτη ερώτηση και μετά όποιος νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει επόμενος. Ε, φυσικά η ερώτησή σας θα έπρεπε να απευθύνεται σε κάποιον εκπρόσωπο της Κομισιόν και να μας πει γιατί τόσο για τα θέματα της Ελλάδας όσο και για τις υπόλοιπες χώρες δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα σε μια χρυσή ευκαιρία για να δείξει η ίδια η Κομισιόν ότι καταλαβαίνει ότι η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης έχει ακριβώς αυτό το ε, ε, έλλειμμα δημοκρατικών, το χαρακτηριστικό έλλειμμα δημοκρατίας που όλοι βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Ε, θέλω να αναφερθώ και στη, λιγάκι στην ε, ερώτηση της ε, κυρίας από τη Γαλλία. Υπάρχει εκτεταμένη ε, πληροφορία στο site μας, στο Save Greek Water και στα αγγλικά, που μπορούμε στη συνέχεια να δείτε λεπτομέρειες και να κουβεντιάσουμε για το άρθρο σας και ό,τι θέλετε. Νομίζω πως είναι ειδικά πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες στη Γαλλία ότι ενώ στην Γαλλία υπάρχει αυτή η μεγάλη τάση επαναδετικοποίησης, όχι μόνο στο Παρίσι, στο Μομπελιέ και στις υπόλοιπε χώρε. Στις χώρες του Νότου Δυστυχώ επιβάλλονται αυτές οι πολιτικές, παρότι είναι κερδοφόρες οι εταιρείε και παρέχουν καλές υπηρεσίες. Και αυτό είναι, ε, πρέπει να ασκηθεί πίεση λοιπόν και από το γαλλικό λαό προς τις δικέ τους κυβερνήσει, ε, για να έχουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Um, just in relation to the σε σχέση τώρα με τους μετρητές. Ε, πρώτα απ' όλα η οδηγία πλαίσιο για το νερό δεν απαιτεί ε, χρεώσεις ε, για το νερό οι δαπάνες, η χρέωση γίνεται βάσει της κατανάλωσης στην Ιρλανδία δεν είχαμε μετρητές το πληρώναμε το νερό μέσω της γενικής φορολογίας ε, και αυτά τα χρήματα κατανέμονται στις τοπικές ε, αρχές που διαχειρίζονται τους υδατινούς σπόρους. Είναι πιο ε, σύγχρονος τρόπος όσον αφορά την κατανάλωση νερού. Στην Ιρλανδία χρησιμοποιούμε 20% κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ οπότε οι μετρητές δεν είναι απαραίτητοι. Δεν θα μειωθεί η κατανάλωση Τώρα σε τοπικό επίπεδο να χρησιμοποιεί κανεί μετρητέ για να ανοιχνεύει διαρροέ, αυτό έχει νόημα διότι βοηθά στην ανείχνευση των διαρροών. Αλλά αν βάλουμε μετρητέ ε, σε κάθε νοικοκυριό, το πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο που εξέτασε ε, αυτό το θέμα, δεν έχω βέβαια κάποιο έγγραφο για να σας δώσω, δείχνει ότι το κόστος συντήρησης των μετρητών ε, και διαχείριση ενό συστήματο τιμολόγηση σε σχέση με αυτού του μετρητέ ουσιαστικά δεν βγάζει τα έξοδά του ουσιαστικά ε, επιβαρύνει την ε, πλήρη ανάκτηση κόστους που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε οι χώρες που έχουν πλήρη ε, συστήματα μετρητών έχουν και τις ε, μεγαλύτερη κατανάλωση νερού ανά νοικοκυριά, Ενώ οι χώρες με λιγότερους μετρητές όπως εμείς στην Ιρλανδία έχουν, ε, παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση. Οπότε η, η σχέση μετρητών και καταναλώσεων δεν βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε επίπεδο νοικοκυριών, αντί για αστικό επίπεδο, δημοτικό επίπεδο, ουσιαστικά αν βάλουμε μετρητέ σε επίπεδο νοικοκυριών, ε, μετατρέπουμε το νερό σε αγαθό και αυτό βοηθά την ιδιωτικοποίηση στο μέλλον. Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, όταν υπάρχουν μετρητέ, ε, φορολογείται κανεί στη Γαλλία για παράδειγμα, βάσει τη κατανάλωση ανά ε, νοικοκυριό. αλλά εσείς ε, προτείνατε να πληρώνουμε το νερό με έναν άλλο τρόπο μέσω των φόρων των γενικών φόρων. Αλλά τι γίνεται αν ο γειτονά μου καταναλώνει ε, πολύ περισσότερο από μένα από ποτίζοντα στον κήπο του τρεις φορές τη μέρα. Και κάνει και 100 ντου την ημέρα. Και ενώ εγώ καταναλώνω λιγότερο, δηλαδή για να είμαι λογική, θα σκεφτόμουν για ποιο λόγο να πληρώνω εγώ τη δική του υπερκατανάλωση ενώ εγώ καταναλώνω πιο λογικά εν συντομία. Ξέρετε, αυτό πάντα είναι κάτι που προκύπτει ως ερώτημα, αλλά όπως είπα, κατά μέσο όρο τα Ιρλανδικά νοικοκυριά καταναλώνουν 20% κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. είναι μύθος το ότι ο κόσμος περνάει μισή ώρα στον ντους ή ότι σπαταλά νερό. Η πλειοψηφία του νερού χρησιμοποιείται στη γεωργία και στη βιομηχανία και αυτοί δεν καλύπτουν την πλήρη ανάκτηση του κόστους δεν έχει λογική το ότι βάζουμε μετρητέ και ο κόσμο έτσι καταναλώνει λιγότερο νερό. Αυτό που δουλεύει είναι εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, όπου διδάσκουμε του ανθρώπου πόσο σημαντικό είναι το νερό και η διατήρησή του και η εξοικονόμησή του. Και αυτό κάνουμε στην Ιρλανδία μέσω ενό συστήματο πράσινη σημαία στα σχολεία και φέρνει αποτελέσματα γιατί στην Ιρλανδία δεν σπαταλάμε νερό. Έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση από τι χώρε που έχουν μετρητέ. επιγραμματικά να απαντήσω λίγο στην ερώτηση του κ. Καρύμπ. Ε, Εμεί, σαν ε, γεωλόγοι, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ένα πηγάδι βρίσκεται μόνο το εκεί πέρα, μια γεώτρηση ή μια πηγή σε ένα άλλο σημείο. Υπάρχει ένα ιδετικό σύστημα, το οποίο ορίζεται μέσα στην οδηγία από τι αποτελείται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση, προφανώ και επειδή έχουν καταγραφεί όλα τα σημεία ύδατο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αν η δικιά σα περιοχή, για παράδειγμα, μπει σε κάποιο μελλοντικό σχέδιο ιδιωτικοποίηση, προφανώ και θα αναγκαστείτε να επιβαρυνθείτε το κόστος που θα ορίσει η εταιρεία η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του νερού. Και θα, πιστεύω ότι αυτό, με βάση τι πρακτικέ που έχουμε, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ανά τον κόσμο, που η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε υποβάθμιση τη ποιότητα του νερού, πιθανώ και με τι μεταλλευτικές δραστηριότητε που αναπτύσσονται στην περιοχή μα στην Ελλάδα, στη, στη πιθανώ πιθανώς στη Φωκίδα ή σε Θάσο που έχουμε τα Μάρμαρα, να έχουμε αποτελέσματα τα οποία μακροπρόθεσμα να είναι αρνητικά και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά τα κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση ε, που πρέπει... Μπορούμε να απαντήσουμε. Ε, ε? Ποιο θα απαντήσει την τελευταία ναι. ερώτηση. Επειδή έχω το κείμενο εδώ που λέει και τι αποφάσει, και μπορεί να μην καθυστερούμε. Ε, καταρχήν το Σύνταγμα τη Ελλάδο με δύο άρθρα. Αναφέρομαι στην, ε, στην ερώτηση που κάνει ο συνάδελφο ο κ. Μαστοράκη. Ε, με δύο άρθρα δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΔΑ και επέκταση των εταιριών ίδρυσης, έτσι. Έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπαριθμό 1906 του 2014 απόφασή τη. Αναλυτικά η Ολομέλεια του ΣΤΕ έκανε δεκτή την αίτηση των κατοίκων τη Αθήνα που ζητούσε να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε χωρί αντάλλαγμα από το ελληνικό δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίηση Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου του λεγόμενου ΤΑΙΠΕΔ το 34% του μετοχικού κεφαλαίου τη ΕΙΔΑΠ. Όπω αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η μετατροπή τη ΕΙΔΑΠ σε ιδιωτική επιχειρήση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματο που επιβάλλουν τη μέρημνα του κράτου για την υγεία των πολιτών αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία τη υγεία. Στην απόφαση αυτή σημειώνεται ότι ο χαρακτήρα τη δημόσια επιχείρηση αναιρείται σε περίπτωση τη αποξενώσεω του ελληνικού δημοσίου από τον έλεγχο τη ΑΕ για του μετοχικού κεφαλαίου ή τη τη αποξενώσεώ του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Εν κατακλείδη, για να μην διαβάσω όλη τη σελίδα, η δικαστική απόφαση επισημαίνει αβεβαιότητα ω προ την παροχή προσιτών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια σε αυτό το βαθμό αναγκαιότητα δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματο, ειδικότερα μετά από το 6 Τετάρτου 2001 ψήφισμα τη 7η Αναθεωρητική Βουλή και κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία τη υγεία, καθώ και στο άρθρο 21 παράγραφο 3 που ορίζει το κράτο μεριμνά για την υγεία των πολιτών. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ε, δεν έχει υλοποιηθεί. Ε, απλά να ολοκληρώσω. Όχι, δεν ναι. Ε, ε, μισό λεπτό. Δεν έχει υλοποιηθεί. Το 27% του μετοχικού κεφαλαίου τη ΕΕ παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ και σκοπεύουν το 27% που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ συν το 34% που είναι στο δημόσιο να μεταφερθεί στο νέο υπερταμείο ιδιωτικοποίησεων. Δηλαδή πάμε σε μια ολική ανατροπή τη εφαρμογή τη απόφαση του ΣΤΕ στην ουσία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει. Να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα και το ενδιαφέρον που δείξατε για τη σημερινή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω του συναδέλφου τον κύριο Εκ, τον κύριο Λόπε και την κυρία Μπόιλεν και του εισηγητέ μα για την ε, παρουσία του εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.